Um, um, λοιπόν, συνάδελφοι, για να εξηγήσω και στα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και σε δεν ήταν εδώ όταν εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη. Προσθέσαμε λοιπόν άλλη μία ψηφοφορία στις ε, ψηφοφορίες ε, συνέστησαν οι συντονιστές σύμφωνα με το άρθρο 99.5 για, το, για την σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης για την Πολωνία πρόταση των Πρασίνων που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τους συντονιστές ζήτησε μια ομάδα στην αρχή της συνεδρίας σύμφωνα με το άρθρο 205 να ψηφίσουμε στην αρχή της ε, ψηφοφορίας για να δούμε εάν ε, εγκρίνονται οι συστάσεις των συντονιστών. Σύμφωνα με το άρθρο 205 μου λένε εδώ πέρα, να δω αν υπάρχει συνένεση δηλαδή, να δω, μου λένε λοιπόν εδώ, αντί να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 205, ε, κάντε λίγο υπομονή, να ψηφίσουμε για το εάν θα ψηφίσουμε. Και αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες ανησυχίες. Λίγη υπομονή. Για το εάν ε, όλοι, ε, αν μπορούσε να λάβει, ε, αν μπορούσαν οι συντονιστές να λάβουν την απόφαση. Οπότε θα ψηφίσουμε για το εάν θα ψηφίσουμε και μετά θα γίνει η ψηφοφορία και τέλος. Οπότε θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτά μου είπαν να σας πω. Λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία, αν τα παρακολουθήσατε, θα ψηφίσουμε για το εάν θα ψηφίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 205, ε, έτσι ώστε αν οι συνάδελφοι θέλουν να αναπεμφθεί το θέμα στους συντονιστές, να γίνει αυτό. Εάν δεν επιστρέψει στους συντονιστές, τότε ψηφίζουμε για το εάν θα εγκρίνουμε την αρχική απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία των συντονιστών. Ε, διαδικασία σε δύο στάδια. Ελπίζω να γίνει ε, συνενετικά. Το δέχεστε, ε, ρωτώ τους συντονιστές. Αντί για την μάζα εδώ των βουλευτών. Ε, μου κάνουν εκεί κάτι νοήματα. Ναι, αυτό μου είπαν όμως ότι έχουμε ως επιλογή. Οι συντονιστέ λοιπόν. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σόφι. Ναι, ναι είναι αυτό. Κάτι εκεί πέρα κάνει με τους ώμους. Εντάξει, αφού δεν μου πετάς πράγματα, καλά είναι. Οι πράσινοι κάτι σαν... Τι να πω, έχετε παραιτηθεί στη μοίρα σας. Εντάξει. Ναι, ναι, ο χρόνος, οκ. να ψηφίσουμε για το αν θα ψηφίσουμε. Πολύ απλά. Θα γίνει τώρα η ψηφοφορία για το εάν θα ψηφίσουμε ή αν θα ξαναπάει στους συντονιστές το θέμα. Με ονομαστική κλίση. Αν πατήσετε το πράσινο κουμπάκι, συμφωνείτε να ψηφίσουμε μετά. Εάν πατήσετε το κόκκινο, ξαναπάει το θέμα στους συντονιστές. Ε, μα ακούστε λίγο. Το πράσινο σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε, το κόκκινο ότι ξαναπάει στους συντονιστές. Άρχεται η ψηφοφορία. Προσοχή, εντάξει, το καταλάβατε. Να το ξαναπώ. Λοιπόν, επειδή τώρα δημιουργήθηκε μία σύγχυση. Α, το κατάλαβατε, εντάξει. Okay. Oh well. So, so you want to go to the vote? Okay, fine. Okay, so right. That was right. Okay, so the vote is closed. So have you changed? Okay. Εντάξει, τι έγινε, για να δούμε. Αλλάξατε άποψη. Και η ομάδα μου λίγο εδώ πέρα μου τα γύρισε. Ε, τώρα πέρασα. Εντάξει, ωραία. Ζητώ συγγνώμη. so... Yeah, I know, I try. Ε, τι να κάνω, προσπάθησα αρχίσανε να βογκάνε όταν άρχισαν να λέω πράσινο και κόκκινο. Οπότε τώρα πάει πίσω στους συντονιστές. Λοιπόν, τέλος. Ηρεμία, συνάδελφοι. Ε, γι' αυτό σας λέω σκόρδο κρεμμύδι. Τι, τι, πώς αλλιώς να τα πω. Μετά, μετά λέτε αμάν αμάν και μετά συμβαίνουν αυτά. Ε, ειλικρινά άρχισαν μερικοί να βογκάνε και να αναστενάζουν. Λοιπόν, πάει πίσω στους ε, συντονιστές και τέλος. Όχι, τότε εγώ ζητώ γραπτή διαδικασία. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένουμε συνεδρίαση των συντονιστών θα καθυστερήσουμε πολύ. Η συζήτηση έχει γίνει. Εγώ θέλω γραπτή διαδικασία αυτή την εβδομάδα. Καλώς. Κύριε Γιούρεκ, το δέχεστε. Ε, κοιτάξτε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας. Ε, καμιά φορά συμβαίνουν αυτά, υπάρχουν και απρόβλεπτα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά να ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα, Α ε, ήταν αναπάντεχο. Μάλιστα, μας βοηθήσατε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σαρτζεντίνη έκανε την πρόταση για την γραπτή διαδικασία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Ωραία, λοιπόν, γραπτή διαδικασία και βλέπουμε. Λοιπόν, πάει στους συντονιστές ούτως ή άλλως. Με γραπτή διαδικασία. Δηλαδή γρήγορη. Ωραία. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη είναι... Συνεργασία Eurojust με την Γεωργία. Η συγκίτρια είναι η κυρία Κάουφμαν. Σιλβί, θέλετε το λόγο, όχι. Πάμε κατευθείαν στην ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Και πέρας. Και δεκτή. 43 υπέρ ε, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Το επόμενο. Απόφαση του Συμβουλίου για να κυρωθεί η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία τόμων ε, σε σχέση με την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τζοζεφ Νάτς είναι ο εισηγητής. Θέλετε τον λόγο, όχι. Μία ψηφοφορία. Άρχεται. Και πέρασε δεκτή με 44 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το επόμενο είναι το πρόγραμμα Περικλής 4. Ε, Ντένις Ντεγιόγκ, είναι ο εισηγητής. Θέλετε τον λόγο, όχι. Ψηφίζουμε. Συμβαστική ένα. άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή Τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή Συμβαστική 2 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 41, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 44 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 4 αρχή ψηφοφορία. Δεκτή. 47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Σαράντα εννέα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 50 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 10. Όχι, 52 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Πάμε στα εκτιμώντα τροπολογία 20 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 21 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. αρχιετή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 23. αρχιετή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 24 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 1 και 26 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Η 28 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Η 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 30 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας και δεκτή 31 αρχιτή ψηφοφορία πέρας δεκτή 32 αρχιτή ψηφοφορία πέρας δεκτή τελική ονομαστική ψηφοφορία να έρχεται Πέρας. Δεκτή με 43 ψήφους υπέρ, καμία κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον Τένις Δε Γιόγκ. The next vote, colleagues, is, um, Η επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση Κόελιο. για την ε, για τον κανονισμό διαλειτουργικότητας. Κάρλος, θέλετε τον λόγο. Μόνο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Είναι μια πρώτη τεράστια μεταρρυθμισή του συστήματος αυτού, όπως βλέπετε υπάρχει μια ψήφος unblock με μία μόνο εξαίρεση. Νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε καλή δουλειά. Ενισχύουμε την ασφάλεια της ζώνης Σέγγεν και προστατεύουμε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κάρλος. Λοιπόν, να δούμε τώρα την προσθήκη, πρώτα την προσθήκη του εισηγητή. Όλους τους συμβασμούς από κοινού, εκτός από τον 7α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 7α. Στη σελίδα 12 του εκλογικού καταλόγου, του καταλόγου ψηφοφορίας, συγγνώμη, 7α. Λοιπόν, 7α, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη σελίδα 44. την τροπολογία 387. Σελίδα 44. Τροπολογία 387. Άρχεται η ψηφοφορία για το 387. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε ούτως ή άλλως. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. 3.93 τώρα. 3.93. Στην ίδια σελίδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τέσσερα στη σελίδα 50. τέσσερα δύο, τρία αρχισε η ψηφοφορια Τέσσερα δύο 3 Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Λοιπόν, από την ομάδα δημοσιονομικών τώρα, τρία, τροπολογία 3, σελίδα 73, τελευταία σελίδα. Τελικά τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία για την τροπολογία 3 της Επιτροπής Τροπολογισμού. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και τώρα τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 30 υπέρ, 8 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την ψηφοφορία. «11 Φεβρουαρίου θα έχουμε μια άλλη συνάντηση στο από τη συνάδελφη.